So uh, the only thing we are voting on is oral amendment number three. Who is in who is in favor? Ψήφι κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά επί της εκθέσεως στο σύνολό της. two Έχουμε δύο απόντες από την ψηφοφορία. Okay. Okay, it's, it's Έγινε δεκτή 19 ψήφοι υπέρ, μηδέν ψήφι κατά, δύο Και τώρα περνάμε στο ψήφισμα. Άρχη ψηφοφορία. And it has been adopted by... Έγινε δεκτό με την αυτή με το αυτό αποτέλεσμα 18 ψήφοι υπέρ, 2 αποχές, καμία αποχή. Περνάμε τώρα στο ε, σημείο 20 που αφορά στην συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες προστασία προσωπικών πληροφοριών ή δεδομένων, πρόληψη, έρευνα και δίωξη ποινικών αδικημάτων. Δια ανατάσσεως της σειρός. παρακαλούμε. Ψηφιπέρ, κατά, Εποχές. δεκτή. Συγχαρητήρια στον κύριο Τζαμπάσκι. Λοιπόν, σημείο 21. Θέμα που αφορά την πρόσβαση στα φάρμακα, εισηγητή ο κύριος Ντουιρόν. Συμβαστική πρόταση ψηφιπέρ Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή απορρίπτεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτέως 46 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ κατά επαλήθευση adopted. Δεκτή. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. αποχέ, Δεκτή. Δεκτό, συγγνώμη. Συμβαστικό σφαιρμός 4 υπέρ. Κατά. αποχέ, δεκτό, 59 τροπολογία υπέρ. Κατά. Επαλήθευση παρακαλώ. It uh, Έγινε δεκτός 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 66 υπέρ κατά αποχές δεκτό, δεκτή 67 υπέρ κατά αποχές δεκτή Συμβασμός 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτός. Συμβασμός 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτός. 76 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμός 7 υπέρ. Κατά. Αποχές Δεκτός. Τροπολογία 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 89 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 91 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση παρακαλώ. έγινε δεκτή. Συμβασμός 8 υπέρ κατά αποχές δεκτός. Τροπολογία 7 ε, υπέρ κατά επαλήθευση. δεκτέ. Ο κύριος Ζεύκα δεν ε, έχει την ε, κάρτα του για να ψηφίσει, οπότε ψηφίζει ανατάσεως ε, τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό συμβασμός 9 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτός, συμβασμός 10 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή 14 υπέρ κατά θα επαληθεύσουμε απορρίπτεται Συμβασμό 11 υπέρ. Κατά. αποχέ δεκτό. 17 τροπολογία υπέρ. Κατά. Νομίζω πως απορρίπτεται, αλλά σε παληθεύσουμε καλού κακού. δεκτής, δεκτός 22 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή 27 υπέρ κατά επαλήθευση. Ναι, 27, 27 τροπολογία. Δεκτή. Τροπολογία 28 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή όπως και το σύνολο του ψηφίσματος το γνωμοδότησης υπέρ κατά αποχές χαρτίρια κύριε Ντυρό η έκθεση σας έγινε δεκτή Uh, Και τώρα έχουμε την έκθεση του κυρίου Χρυσόγονου, αριθμός 22, αρχίζει η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. So this has been clearly adopted. Congratulations to Mr. Συγχαρητήρια τον κύριο Χρυσόγων. Έγινε δεκτό το θέμα 22. Το 23 έχει αναβληθεί, έχει μετατεθεί. So that's all for the vote. Uh, now let me, let me... Αυτά σε ό,τι φορά τις ολοκληρώσαμε. Τώρα περνάμε στις ε, δηλώσεις Προέδρου σχετικά με ε, τη συζήτηση στο πλαίσιο των συντονιστών. Ε, έγιναν δεκτή, δεκτά τα ονόματα των εισηγητών, ο κ. Καβαντά και η κυρία Για το ζήτημα των έργων τέχνης, εγώ ο υποφαινόμενος ε, Ασυρία του κυρίου Μαρίνιο Πίντου, ο κύριος Λεμπρετό, ασυλία της κυρίας Λεπέν, με κυρία Φεράρα, η συγγήτρια και το χρονοδιάγραμμα είναι δεκτό για το 2017 χωρίς αλλαγές. Τρίτον, ο κ. Ζεύκα ορίστηκε ως μέλος ε, του δικτύου αναφορών Οι συντονιστές συμφώνησαν ε, να υποβάλουν γραπτή ερώτηση σχετικά με την ε, θέμα των εγγράφων. Αυτό το θέμα θα ακολουθήσει την γραπτή διαδικασία. Σημείο 5. Ε, τον Ιστέ ζήτησαν από την Γραμματεία να ετοιμάσει μια έκθεση για μια γνώμη για την ε, θέμα του Brexit. Ε, συμφωνήσαμε να καλέσουμε τον πρόεδρο Μπατιστέλη και τον, πρόεδρο, τον που να μας μιλήσει τον Ιανουάριο 2017 μαζί με τον κύριο Λένε και τον κύριο Μπαλτασάρη και τον κύριο Ραπκάι. Οι συντονιστές αποφάσισαν να ε, διοργανώσουν μια εκδήλωση με την Επιτροπή ΕΦΚΟ για την 60η επέτειο ε, από την ε, συνθήκη της Ρώμης. Οι συντονιστές έλαβαν γνώση ένα ψήφισμα και αποφάσισαν να μην αναλάβουν περαιτέρω δράση. Τέλος, οι συντονιστές αποφάσισαν να καλέσουν τον κύριο και πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου, τον 2017 ε, για ανταλλαγή απόψεων. Αυτές είναι αποφάσεις λοιπόν των συντονιστών και μπορούμε να συνεχίσουμε με το υπαριθμόν 24 ζήτημα. Ανταλλαγή απόψεων για την τροπολογική οδηγία 2004-37 για την προστασία των εργαζόμενων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες ή μεταλλαξιογόνες ουσίες. Το λόγο έχει ο κύριος Χρυσόγωνος. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ο καρκίνος είναι η βασική αιτία θανάτων που σχετίζονται με την εργασία, ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Ο, ο καρκίνος όχι μόνο ε, μειώνει την ε, ποιότητα ζωής, αλλά έχει σαν αποτέλεσμα αύξηση κόστους άμεσα και έμεσα ο καρκίνος έχει επίσης ε, αρνητικές επιπτώσεις σε όλη την κοινωνία γιατί μειώνει την παραγωγικότητα και αυξάνει το, τις δημόσιες ε, δαπάνες και ο καρδιός θέεται με την θέση εργασίας, ε, συνεπάγεται αύξηση κόστους για την ανάγκη αντικατάσταση των εργαζομένων και επίσης ε, αύξηση κόστους σχέση με την παροχή αποζημιώσεων. Η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η τροποποίηση της ε, οδηγίας για την προστασία των εργαζομένων όσον αφορά τους κινδύνους που προέρχονται από καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες ουσίες στο χώρο εργασίας έχει σαν στόχο να μειώσει τον κίνδυνο έκθεσης σε τέτοιου είδους ε, καρκινογόνες ε, ουσίες, να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της ελωσιακής νομοθεσίας στον τομέα αυτό και να παράσχει μεγαλύτερη σαφήνεια και καλύτερους όρους για όλους τους οικονομικούς παράγοντες. Αυτή η πρόταση έχει σαν στόχο να συμπεριλάβει στο πεδίο, οδηγίας, ε, στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας έναν κατάλογο χημικών ουσιών Monomer respirable crystalline silica dust, hydrazine. Ε, διάφορες ε, ουσίες ρητίνες ε, κλπ. που αναγνωρίζονται ως ε, ε, καρκινογόνες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από διεθνείς οργανισμούς όπως είναι ο Διεθνής Οργανισμός για την Έρευνα του Καρκίνου αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν ταξινομηθεί εντός του τρέχοντος ευρωπαϊκού συστήματος. Η πρόταση επίσης έχει σαν στόχο να ορίσει κάποιες οριακές τιμές στη βάση των πιο πρόσφατων επιστημονικών ε, τεκμηρίων, εναρμονίζοντας ε, λοιπόν τις ε, εθνικές τιμές, οριακές τιμές εκεί όπου υπάρχουν. με τον τρόπο αυτό θα σωθούν 100.000 ανθρώπινες ζωές το μελλοντικά. Γι' αυτό υποστηρίζω όλες τις τροπολογίες οι οποίες υπογραμμίζουν την ανάγκη να υπάρχει μια πρώιμη παρέμβαση εκεί όπου υπάρχει ανάγκη να αντιμετωπιστούν αυτά τα εξαιρετικά τοξικά μείγματα στα οποία εκτίθενται οι εργαζόμενοι και εκεί όπου δεν υπάρχουν επαρκή μέχρι στιγμής επιστημονικά στοιχεία. Ε, για ένα αποτελεσματικό μοντέλο πρόληψης και αντιμετώπισης του κινδύνου, το οποίο λαμβάνει υπόψη τις ε, διάφορες παραμέτρους που οδηγούν στην ανάπτυξη της νόσου. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να υπάρχουν καλύτερες προδιαγραφές υγείας για τους εργαζόμενους και να ανταπιστούν Καταστάσει που αφορούν ακριβώ την έκθεση των εργαζομένων και προκειμένου να διαφυλαχθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα ε, υγείας ε, ε, και εργασία. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μαρίνο Πίντο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ μπορώ να υποστηρίξω την πρόταση του ΣΥγητή και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ήθελα να εκφράσω και μία ιδέα. Επί χρόνια, επί δεκαετίες, το αίτιο του καρκίνου ε, θεωρείται ότι οφειλόταν βασικά σε γενετικά προβλήματα. Και τώρα έδειξε η επιστήμη ότι υπάρχουν και συγκεκριμένα αίτια από την έκθεση σε κάποια προϊόντα που δημιουργούν καρκίνο. ή κάποιες συνθήκες εργασίας οδηγούν σε καρκίνο. Έτσι, πολλές επιθετικές μορφές καρκίνου είναι αποτέλεσμα Ελήψεως σωστών συνθήκων στο χώρο εργασίας. Είναι επαγγελματικέ ασθένειες. Άρα χρειάζεται ε, να γίνουν νομοθετικές αλλαγές για να αποζημιωθούν τα θύματα για αυτή την κατάσταση. Πολύ συχνά βλέπετε όλα αυτά οφείλονται σε αμέλεια των εργοδοτών αλλά και στην έλλειψη επενδύσεων, σαφή έλλειψη επενδύσεων για να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και να δουλεύει ο άνθρωπος σε υγιεινές συνθήκες και να αποφεύγει αυτές τις ασθένειες, διάφορες ασθένειες μεταξύ των οποίων και ο καρκίνος, που ο καρκίνος είναι βασική επαγγελματική ασθένεια. Λοιπόν, ε, χαίρομαι υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία και σίγουρα θα πρέπει να εγκριθεί στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ζητάει άλλο το λόγο για αυτό το θέμα. Όσον αφορά τώρα το όλο πρόγραμμα, ο κ. κύριε Χρυσόγωνε, είναι αυτό που αναφέρεται. Ωραία. Δεν αλλάζει τίποτα. Όπως φαίνεται στο, στο έγγραφο. το το για τροπολογίες κλπ. Εφόσον είσαστε εδώ παρόν κύριε Χρυσόγωνε, Μήπως μπορούμε να πάρουμε το σημείο που δεν συζητήσαμε χτες, το απόγευμα. Το σημείο 31, με άλλα λόγια. Έτσι, εν συντομία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2008-52 για κάποιες πτυχές διαμεσολάβησης σε εμπορικά και αστικά θέματα. Η Οδηγία 2008 κάθετος 52 για κάποιες πτυχέ διαμεσολάβησης σε θέματα εμπορικά και αστικά εφαρμόζεται σε διασυνοριακές διαφορές όσον αφορά αστικά και εμπορικά ζητήματα καθώς και στο τομέα του οικογενειακού δικαίου. Αυτή η οδηγία προσπαθεί να διευκολύνει την πρόσβαση σε εναλλακτικέ διευθετήσεις των διαφορών και να προωθηθούν οι φιλικέ διευθετήσει των διαφορών τη χρήση της διαμεσολάβησης εξασφαλίζοντας σωστές σχέσεις μεταξύ διαμεσολάβησης και δικαστικών α, και εκδικάσεως υποθέσεων. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η διαμεσολάβηση μπορεί να είναι αποτελεσματική όσον αφορά το κόστος και με εξώδικη επίλυση των διαφορών σε αστικά και εμπορικά θέματα μέσω διαδικασιών που ταιριάζουν στις ανάγκες των μερών και έτσι τα μέρη πιο πολύ θα μπορέσουν να προσφύγουν σε συμφωνίες μέσω διαμεσολάβησης. Η διαμεσολάβηση είναι χρήσιμο εργαλείο παρέχει αυξανόμενη πρόσβαση στη δικαιοσύνη και ελαφραίνει το άχθος ε, όσον αφορά το δικαστικό σύστημα που ήδη έχει μεγάλο βάρος. Μέσω επικαιροποιημένη μελέτη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γενική Διευθύνσεω για τα θέματα δικαιοσύνη και καταναλωτών και περαιτέρω στοιχεία, εμφανίζεται ότι η εφαρμογή τη οδηγία για τη μεσολάβηση είχε σημαντικό αντίκτυπο όσον αφορά την νομοθεσία διαφόρων κρατών μελών πέρα από την θέσπιση κάποιων προαπαιτούμενων για τη χρήση διαμεσολάβησης διασυνοριακές διαφορές για τα εμπορικά και αστικά θέματα. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η οδηγία έχει προωθήσει τη διαμεσολάβηση και σε εσωτερικές διαφορές ε, εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν επεκτείνει το πεδίο των μετρών, μέτρων τους εφαρμόζοντας την οδηγία και σε εσωτερικές υποθέσεις, όχι μόνο τις συνοριακές. Σαν αποτέλεσμα η οδηγία έχει δώσει προστιθέμενη αξία στην Ευρωπα... της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ευαισθητοποιώντας τους εθνικούς νομοθέτες όσον αφορά τα ωφέλη της διαμεσολάβησης. Απ' την άλλη πλευρά, δυσκολίες που αφορούν τη λειτουργία των εθνικών συστημάτων διαμεσολάβησης στην πράξη σχετίζονται βασικά με την, αντι... την ε, τη... τη συγκρουσιακή προσέγγιση που ακολουθούν τα κράτη-μέλη και την, ε, την έλλειψη ελεκτικών μηχανισμών και τα μέτρα που είχαν χρησιμοποιηθεί για την πρόθεση της διαμεσολάβησης και την εκπαίδευση του προσωπικού δεν επεκτείνουν τη χρήση της διαμεσολάβησης όσο ταχαίως ε, ε, ελπίζαμε. Η χρήση της διαμεσολάβησης ε, οδηγεί σε πολύ επιτυχία αποτελέσματα. Όμως χρησιμοποιείται σπάνια συστηματικά η διαμεσολάβηση από τους εμπλεκομένους φορείς και τους νομικούς και τους διαδίκους. Δεν χρειάζεται να θέσει οδηγίε σε αυτή τη φάση. Όμω η εφαρμογή της θα πρέπει να βελτιωθεί και αυτό να γίνει μέσω μέτρων. Επειδή είναι πολύ επιτυχή η διαμεσολάβηση, δεν χρησιμοποιείται αρκετά, πρέπει να γίνει η διαδικασία ευαισθητοποίησης, να μάθει το κοινό την ύπαρξή τη και πόσο χρήσιμη είναι. Η διαμεσολάβηση, βλέπετε, δεν χρησιμοποιείται παραδοσιακά στη θέση των διαφορών, Γι' αυτό πρέπει να δοθούν κίνητρα να χρησιμοποιείται. Και πάνω απ' όλα είναι σημαντικό να αποδειχθεί ότι δίνει ωφέλη η διαμεσολάβηση. Και θα πρέπει έτσι να εφαρμόζεται η οδηγία του 2008 για τη μεσολάβηση. Η προθεσμία υποβολή τροπολογιών είναι 8 Φεβρουαρίου του 2017. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αν επιτρέπετε, να σας πω το εξής. Όσον αφορά αυτό το θέμα, θα διεξαχθεί ένα εργαστήριο στις 29 Νοεμβρίου από τις 4.30 μέχρι τις 6.30 το απόγευμα. Ευχαριστώ. Δεν ζητά κάποιος το λόγο, άρα μπορούμε να συνεχίσουμε και να πάμε στο σημείο 26 νομίζω. 26 σχέδιο γνωμοδότησης για τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Καναδά όσον αφορά την εφαρμογή της δικής τους νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. Η συγγητής ο κ. Λεμπρετών. Έχετε το λόγο κύριε Λεμπρετών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το εμπόριο ανάμεσα στην Ένωση και τον Καναδά καλώς έχει από το 1999 εφίσταται συμφωνία ανάμεσα στα δύο μέρη που βασίζεται στην συνεργασία ανάμεσα στις ε, αρχές ανταγωνισμού και είναι μια συμφωνία η οποία έχει δείξει την σημασία της ε, εδώ και 17 χρόνια και αυτό προς ικανοποίηση των πάντων. Ε, θέλαμε λοιπόν να επικαιροποιηθεί και αυτό είναι το αντικείμενο του κειμένου του θα γνωμοδοτήσουμε σήμερα διευκρινίζω πως δεν έχει καμία σχέση με την συμφωνία ΣΕΤΑ. Πρόκειται για κάτι τελείως διαφορετικό. Αντικείμενο αυτής τη βελτίωσης είναι η διευκόλυνση τη ανταλλαγή ε, της ανταλλαγής ε, πληροφοριών ανάμεσα στις ε, αρμόδιες περί ανταγωνισμού αρχές, έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν τι κάνουν οι μεν και οι δε. Η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών είναι εγγυημένη. Τώρα, τακτικέ συναντήσει ανάμεσα στα μέρη θα ε, οργανωθούν για την βελτίωση αυτών των πληροφοριών και των ανταλλαγών. Πρόκειται για μια συμφωνία καθαρά τεχνικού χαρακτήρα, η οποία χρειάζεται να βελτιωθεί. Άρα είμαι υπέρ. Εκφράζομαι λοιπόν υπέρ. Εντάξει, δεν επιθυμεί κάποιο να απαντήσει. Να πω ότι οι προθεσμίε για την ε, υποβολή τροπολογιών είναι 11 ε, Νοεμβρίου το μεσημέρι τροπολογίες ε, γίνονται παραδεκτές ε, εάν ακολουθούν την σύσταση του εισηγητή και υπενθυμίζω ότι η ψηφοφορία δεν μπορεί να διεξαχθεί προτού να μας ζητηθεί επισήμως από το Συμβούλιο. να καλωσορίσω την αντιπροσωπεία της οργάνωσης Χαλκίτα Μπαρ της Ίσως πρόκειται για την Ένωση Δικηγόρων Χαλκίδας. Περνάμε στο σημείο 8 ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την απαλλαγή του 2015 και το λόγο έχει εκ νέου ο κύριος ε, Λεμπρετό. Και εδώ λοιπόν ε, εκφράζω θετική γνώμη για αυτή την απαλλαγή διότι υπάρχουν ε, πολλά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να πιστωθούν υπέρ του δικαστηρίου το πρώτο στοιχείο είναι ότι το ελεγκτικό συνέδριο δεν, ε, δεν έκανε δικές ε, απαντήσεις αναφορικά με την λειτουργία του δικαστηρίου. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι οι στατιστικές είναι αρκετά καλές, ικανοποιητικές, διότι η διάρκεια των διαδικασιών του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι 15 μήνες για τις προδικαστικά, 17 μήνες για τις ε, υπόλοιπες περιπτώσεις. Τώρα σε ό,τι φορά το δικαστήριο η διαδικασία είναι 20 μήνες και μισό και για το δημόσιο, για δικαστήριο για τα δημόσια ζητήματα είναι, 20, είναι 18 μήνες τώρα. Οι αποφάσεις ήταν σε αύξηση σε σχέση με το παρελθόν, πρόκειται για 4% επιπλέον υποθέσεις που έχουν εξεταστεί. Το τέταρτο στοιχείο ευνοϊκό είναι ότι η εφαρμογή, η κούρια, δηλαδή η δυνατότητα της ανάθεσης ε, με ηλεκτρονικά και αυτή έχει αυξηθεί σημαντικά. Το 2009 ήταν 114 ε, ενώ 230 το 2014 και το πέμπτο και τελευταίο στοιχείο το οποίο είναι ευνοϊκό, υπέρ δηλαδή του δικαστηρίου, ότι η ισορροπία ανάμεσα σε άνδρες γυναίκες για θέσεις ευθύνης και εδώ έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Άρα δεν υπάρχουν παρά μόνο θετικέ εξελίξει, κάτι το οποίο με οδηγεί στο να γνωμοδοτήσει υπέρ τη απαλλαγή. Ευχαριστώ. κύριο κύριο Ζιεφκά έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λεμπρετό για την, την ε, σύντομη παρουσίαση Λυπούμε που πολλοί συνάδελφοι απουσιάζουν κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων μας, ιδιαίτερα τα άτομα τα οποία ήταν κατά τη μεταρρύθμισης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Τα δεδομένα που μας παρουσίασε ο εισηγητής καταδεικνύουν ότι πόσο απαραίτητη ήταν αυτή η μεταρρύθμιση και πώς πήγε προς σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, μάλλον αυξάνονται συνεχώς οι περιπτώσεις που εξετάζει το δικαστήριο και άρα θα πρέπει να αυξηθεί και ο αριθμός των δικαστών. Ακόμα και ο χρόνος ε, μέσα στον οποίο εξετάζονται οι υποθέσεις έχει περιοριστεί. Αλλά παραμένει κατ' εμέ αρκετά υψηλό αυτό το διάστημα. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται περισσότερους δικαστές. Έχουμε βελτιώσεις λοιπόν σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος ε, αυτό χάρη στις προφορίες ε, που λάβαμε από το ελεγκτικό συνέδριο μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι οι μεταρρυθμίσεις ε, εφαρμόζονται σωστά στο δικαστήριο και όπως γνωρίζουμε τα πάντα θα αναλυθούν μέσα σε κάποια χρόνια. Αλλά ακόμα και τώρα, αν ρίξουμε μια ματιά στην εικόνα που μας έδωσε ο εισηγητής, έχουμε θετικά συμπεράσματα. Μπορούμε να ολοκλώσουμε λοιπόν αυτό το θέμα, παρατηρεί ο Πρόεδρος. Περνάμε στο σημείο 27. Έλεγχος ε, εφαρμοστικών πράξεων και ε, αυτό αφορά τους κανονισμούς της ε, Κομισιόν και σε σχέση με τον κανονισμό 655 2014 Δυστυχώς ε, δεν έχουμε τον εισηγήτρια κυρία Φεράρα, αλλά δεν έχει αντιρρήσεις ε, πάνω στο θέμα, δεν έχει στάσεις, ε, εκτός εάν έχουν οι παρόντες. Αν δεν υπάρχουν στάσεις μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση επί του ζητήματος αυτού. Και αυτό ήταν το τελευταίο θέμα μας για σήμερα το πρωί. Να σας υπενθυμίσω ότι το απόγευμα έχουμε το εργαστήριο σχετικά με την αναδιατύπωση του κανονισμού των Βρυξελών. Ευχαριστώ την παρουσία σας σήμερα. Το πρωί